Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Μπάλτσε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ως εισηγητής χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στην ε, συζήτηση μπορούμε να έχουμε τη συμμετοχή του Επιτρόπου. Η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη με μεγάλη πλειοψηφία ότι η νομοθεσία των προηγούμενων πέντε ετών πρέπει να εξεταστεί ε, διεξοδικά. Δεν σημαίνει αυτό απορρίθμιση ε, σημαίνει ότι πρώτα θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό ε, στη, της νομοθεσίας ε, των χρηματοδοτικών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει έτσι να εντοπίσουμε και να άρουμε αδυναμίες. Σημαίνει αυτό επίσης ότι τα αποτελέσματα της, των διαφόρων ρυθμίσεων θα πρέπει να ε, αναδεικνύονται με τρόπο σαφή. Την περίοδο 2007-2008, όταν άρχισε η κρίση, ε, το νομοθετικό έργο δεν είχε ε, αρχίσει. Ε, αρχίσαμε να παίρνουμε μέτρα μεσούσης της κρίσης. Ε, βεβαίως δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Όλο το οικοδόμημα άλλαξε με νέες εποπτικές αρχές, με πρότυπα υποχρεωτικά πανευρωπαϊκά και με την Τραπεζική Ένωση. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε, πρέπει όμως να εντοπίζουμε κενά, αδυναμίες, ασάφειες, ε, υπερβολές. Ε, ως ε, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να κάνει μία μελέτη ε, που θα καλύπτει όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς. Θέλουμε να εξεταστεί ιδιαίτερα τα επόμενα σημεία. Πρώτον, ε, η προσαρμοστικότητα των υπαρχόντων κανόνων και νόμων, γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχουν αμφισημίες ε, και αντιφάσεις. Θα πρέπει να είναι πρακτική η νομοθεσία, να μπορεί να εφαρμόζεται. Ε, Επίση, ε, θέλουμε για τους ε, καταναλωτές να διατηρήσουμε την ε, ε, διαφορετικότητα της αγοράς. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να επιβαρύνουμε πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, η συνθετότητα και η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων που υπάρχουν. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας σε χρηματοπιστωτικά θέματα. Και βέβαια, όταν ε, στο, όταν ε, λαμβάνονται ε, αποφάσεις στη Βασιλεία ή στο Ιώσκο, στη Μαδρίτη θα πρέπει να συμμετέχουμε καθοριστικά. Αυτό είναι σημαντικό και για τους επενδυτές. Ε, δεν θέλουμε να ε, παράγεται μόνο ενημερωτικό υλικό γενικότερα, αλλά υλικό το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των επενδυτών ε, παραγωγών. να μειώνουμε τα εμπόδια και να ε, ανοίγουμε την εσωτερική αγορά στις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες. Τέλος, ε, τα οικονομικά αποτελέσματα, ο οικονομικός αντίκτυπος. Ε, πιστεύουμε ότι η οικονομία είναι ισχυρή εκεί που μπορεί να είναι αποτελεσματική, στην πραγματική οικονομία. γι' αυτό θα πρέπει να δώσει η νομοθέτης τις δυνατότητες. για, για μένα, ως εισηγητή και για το ΕΛΚ, Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να μην αποδυναμωθούν. Χρειαζόμαστε και ζητούμε γι' αυτό μια ανάλυση ποσοτική και ποιοτική από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Η ρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα είναι ο στόχος, ε, όπως και η ε, θα πρέπει να εξασφαλίζει σταθερότητα και να προωθεί τους βασικούς μας στόχους. Ε, ε, ε και για την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική, ε, το χρηματοοικονομικό τομέα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ε, αν θέλουμε να αναζωογονήσουμε τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, νομίζω ότι σε ένα χρόνο, όταν θα συναντηθούμε το... και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, θέλουμε να υπάρχει η μελέτη που ζητήσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Χίλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω ενώπιον σα απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Μπάλτ για την τόσο σημαντική του έκθεση που καταδεικνύεται δικαιωμένα τόσο σαφώ. Σημερίζομαι 100% το στόχο του να υπάρξει ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμω, Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει να ξέρουν περαιτέρω ότι θα έχει αναλογικό χαρακτήρα και ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ερευστέ και πεταλασσόμενε καταστάσει. Αυτή είναι η λογική που διατρέχει <clears throat> την προσπάθεια συλλογή στοιχείων που βρίσκεται πίσω από το σχέδιο δράση για τι αγορέ κεφαλαίων. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση για συλλογή στοιχείων είναι συμβατή με του στόχου. μας. Θέλω να σταθώ τώρα σε δύο θέματα που γύρονται από την έκθεση, την ανάγκη να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. <clears throat> είναι φανερό ότι οι μεταρρυθμίσει που εισαγάγαμε τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τώρα είναι καιρό να δούμε κατά πόσο αυτά τα, 40 νομοθετήματα που έχουμε εγκρίνει είχαν κάποιες απροσδόκητες ε, συνέπειες. Όπως είπε ο κ. Μπάρτς, πρέπει πράγματι να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες μας κάνουν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουν. Αυτή η συλλογή στοιχείων, η πρόσκληση για παροχή στοιχείων θα τελειώσει αυτό το μήνα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει την ε, προσέγγιση μας να <clears throat> εξασφαλίσει μια σωστή αξιολόγηση όλων αυτών των νομοθετημάτων που προβλέπεται να γίνει τα επόμενα χρόνια και θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο εμεί παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα τη νομοθεσία στο μέλλον και η έκθεσή σα έχει μερικέ πάρα πολύ ενδιαφέρουσε σχετικά προτάσει. Χρειαζόμαστε νομοθεσία που έχει αναλογικό χαρακτήρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει την επένδυση. Αν μπορούμε λοιπόν να απλοποιήσουμε και να ευθυγραμμίσουμε την νομοθεσία και παρόλα αυτά να επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο, τότε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. <clears throat> Είμαι έτοιμος να επανέλθω και να σας δώσω αναφορά για τα θέματα αυτά όταν έχει τελειώσει η πρόσκληση για συλλογή στοιχείων το να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων είναι κάτι που υποστηρίζω ιδιαίτερα επίση στην εκθέση του κ. Μπάλτ. Αν θέλουμε οι εταιρείε να μπορούν να ξεκινούν, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν θέσει απασχόληση στην Ευρώπη, θα πρέπει να βελτιώσουμε την δυνατότητα χρηματοδότησή του. Αυτό βρίσκεται πίσω από την πρόθεσή μα να εδραιώσουμε μια αγορά ε, αγορών και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ξέρετε ότι έχουμε προτείνει μια σειρά από την οδηγία για το προσπέκτο, στο διαφημιστικό φυλάδιο δηλαδή, και έχουμε και την πρότασή μα να έχουμε μια διαδικασία τυπλοποίηση που είναι απλή και τυποποιημένη. Αυτό θα βελτιώσει τη δυνατότητα χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα και τη χρηματοδότηση του γενικού οικονομικού χώρου. Το Συμβούλιο λοιπόν έχει φτάσει σε μια κοινή θέση και ελπίζω και το Κοινοβούλιο θα πράξει το ίδιο. Αυτά είναι τα κύρια θέματα που αναφέρονται στην έκθεση Μπάλτσα, αλλά υπάρχουν και πολλέ άλλε προτάσει. Όλα αυτά έχουν ενισχύσει την πεποίθησή μου ότι με το να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε από κοινού έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να βελτιώσουμε την νομοθεσία μας, να εξασφαλίσουμε ότι έχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της παροχής εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και της υποστήριξης επενδύσεων και ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Λεβεντόφσκι, να ο Πρόεδρε, Επίτροπε, είναι φυσικό ε, εν το μέσο της ε, κρίσης που ξεκίνησε ως ε, οικονομική κρίση ε, να αναζητούμε τους κατάλληλους κανόνες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μακροοικονομική σταθερότητα στο μέλλον. Αυτό σημαίνει κόστος και πιο περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον. Ε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε σε ένα βαθμό τις, ε, ε, μη, τα μη τραπεζικά χρηματοδοτικά ιδρύματα. Το, η πράσινη βήλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Χρηματαγορών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ταυτόχρονα ε, το διεθνές περιβάλλον. Γιατί υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον για την πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη συγχρηματοδότηση. Ε, και θα πρέπει να καταργήσουμε και τους φραγμούς αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στον κύριο Μπάλτς και σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 7 χρόνια υιοθετήσαμε ένα μεγάλο αριθμό ε, κειμένων σχετικών με τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όλα σχετικά με την κρίση. Και με αυτόν τον τρόπο ανακτήσαμε και διατηρήσαμε την μακροοικονομική σταθερότητα. Και νομίζω ότι θα αποφύγουμε αυτόν τον τρόπο τις υπερβάσεις ε, και, εν πάση περιπτώσει, θα αποφύγουμε οι φορολογούμενοι να καλύπτουν τέτοιου είδου ε, υπερβάσεις και καταχρήσεις στο μέλλον με τους φόρους που πληρώνουν. Ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τώρα όλο αυτό το πλαίσιο και να δούμε πού πρέπει να διορθωθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό που περισσότερο μου αρέσει στην έκθεση είναι ότι αυτή προτείνει τρόπους για την μέτρηση της πρόσβασης που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε χρηματοδότηση επίσης στην μέτρηση των ε, εμποδίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάγκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα δεν πάει καλά, δεν είναι αρκετέ οι επενδύσει, οι τράπεζε δεν ανταποκρίνονται, οι κεφαλαίοι αγορέ δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώ. Η Ένωση Κεφαλαίου λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μια δυνατότητα για χρηματοπιστωτικές, χρηματοοικονομικές καινοτομίες. Οι φραγμοί μεταξύ κρατών μελών μπορούν έτσι να ξεπεραστούν και η Επιτροπή ε, μελέτησε το σύστημα στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου εκεί το 80% ε, των ε, δανείων δίνονται από τις κεφαλαγορές. Εδώ το 20%. Ε, δεν είμαστε Ηνωμένε Πολιτείε, όμως πρέπει να, να αναπτυχθούν οι κεφαλαίοι αγορές, αλλά θα πρέπει και οι δημοσιονομικές ε, υπηρεσίες να ρυθμίζονται καλύτερα και οι διαδικασίες. Αν δούμε στις, τις ΗΠΑ, εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ αποταμιεύσεων και ε, τραπεζικών επιχειρηματικών εργασιών κτλ. Η έκθεση ε, παίρνει ως βάση έναν ε, ε, τομέα που θα εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία. Η απορρίθμιση θα είναι μόνο ε, μέσον, όχι αυτός σκοπός. Είναι ισορροπημένη η, έκθεση, η προσέγγιση αυτή. άρα μπορούμε και εμείς να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Πρέπει όμως ο χρηματοπιστωτικός τομέας να ειδωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να αποδίδει, να προσφέρει υπηρεσίες. Η κεφαλαία αγορά μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν αναγνωριστεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να δώσουμε έμφαση στις ε, επενδύσεις, ε, στις καινοτομίες, μόνο έτσι θα υπάρξει ανάπτυξη. Η κυρία Σουίνμπορντ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά για του εισηγητή και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προέβησε σε πολλά νομοθετήματα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε τα κενά της επικαλύψης. Η έκθεση αυτή του κυρίου Μπάλτσε λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε ε, πέρα από δηλώσεις ε, αρχών. Θα πρέπει να δούμε και συγκεκριμένες ποσότητες. Ε, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία επικάλυψη κυρίως ε, μεταξύ νομοθετημάτων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, και το CND4 και το MIFID κυρίως. Θα πρέπει λοιπόν να τα λύσουμε αυτά. Επίσης θα πρέπει να δούμε την υποχρέωση συμψηφισμών. Ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, έπρεπε να περιοριστούν σε ε, ορισμένου, ώστε να μην υπάρχουν αθέμητες ε, πρακτικές. Αυτό όμως δημιούργησε υπερβολικό, υπερβολικό φόρτο στη λειτουργία τους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιέζεκ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαίρομαι για το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής της έκθεσης είναι σημαντικό να προχωρήσουμε από την δημιουργία νέας νομοθεσίας στο να κλείσουμε τα κενά και να βελτιώσουμε τις ατέλειες της ε, υπάρχουσας νομοθεσίας για να υπάρξει μεγαλύτερη ενθάρρυνση για την επένδυση στην Ευρώπη. Ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης απολογισμού είναι να μπορέσει η Κομισιό να κάνει ένα συνολικό απολογισμό των ε, νομοθετικών πράξεων και με τον τρόπο αυτό να εξετάσει όλες τις νομοθετικές πράξεις που έχουν εφαρμοστεί με την χρηματοπιστωτική κράση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η έκθεση αντικτύπου και αξιολόγησης να δει πώς τα διάφορα τμήματα της νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αλληλεπιδρών. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν παραθυράκια, υπάρχουν συνέπειες που δεν έχουν προβλεφθεί είναι κάτι το οποίο έχει βλάψει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης συνολικά. Θα πρέπει να αποκτήσουμε μια πλήρη κατανόηση της νέας νομοθεσίας αυτής για να μπορούμε στη συνέχεια να εργαστούμε καλύτερα για να φτιάξουμε ένα πιο ανθεκτικό και πλήρε σύστημα για κεφαλογικές αγορές. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό σημαίνει θα πρέπει να έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες. Τρίτον, θα πρέπει να δώσουμε την καλύτερη πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κεφάλαια για να υπάρχει μόνιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ρυθμιστική διαδικασία δεν <clears throat> τροχοπεδεί αυτή τη διαδικασία και να μειώσουμε το άχθος για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν να κάνουμε με υπερβολική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεμάση έχει το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την απορρίθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται υπό το πρόσχημα της λεγόμενης καλύτερης νομοθεσίας. Αλλά μια ευφύης ρύθμιση της, ε, των χρηματοπιστωτικών θεμάτων δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη. Η δική μου νομοθεσία έχει χίλιε σελίδε για μια νομοθεσία η οποία καλύπτεται στι ΗΠΑ από 37 σελίδε. Έχουμε πολλές ε, τράπεζε οι οποίε είναι υπερβολικά ισχυρέ και αυτό δεν έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό των τραπεζών που είναι too big to fail. Η σωστή άποψη που δεν επεκράτησε ήταν να κοπούν σε κομμάτια αυτές τις τράπεζες, να διαλυθούν σε τμήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δίνει την εντύπωση ότι θα μπορέσει με την συνθετική τυπλοποίηση να λύσει το πρόβλημα χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που φταίει όμως είναι η πολιτική λιτότητα και η αδυναμία να εξετάσουμε καλύτερα τους τραπεζικούς ισολογισμούς και τα κενά που έχουν. Το παραμύθι λοιπόν αυτό ότι θα κερδίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή τη διαδικασία είναι ένα παραμύθι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να έχει περισσότερες τράπεζες οι οποίες πρέπει να βρίσκονται κάτω από δημόσιο, έργο, δημόσιο έλεγχο και καλύτερο έλεγχο του τραπεζικού τομέα. Η μόνη πραγματική καινοτομία που έχει γίνει στον τομέα αυτό είναι τα ATM. Ο κύριος Γκίγκολτ έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφε Μπάλτς, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν η έκθεση αυτή ε, βάζει τις σωστές προτεραιότητες. Η κυρία Σουίνμπουρ είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε έκκληση για μονοπλευρή απορρίθμιση. Διπλή απορρίθμιση αλλά και κάλυψη των κενών, μείωση της ε, περιπλοκότητας που είναι άχρηστη αλλά όχι μονοπλευρή απορρίθμιση. Το λέω αυτό για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Τονίζεται σωστά ότι στην έκθεση ότι σε ορισμένους τομείς δεν κάναμε αρκετά. Σε άλλους δεν προχωρήσαμε με βάση την αναλογικότητα. Αυτό στην ε, ε, νέα επεξεργασία θα παίξει ρόλο. Επίσης, ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει να το δούμε μέσα από το πρίσμα του χρήστη. Ε, κάποια χρηματοπιστωτικά προϊόντα είναι δηλαδή ιδιαίτερα ακριβά σε σχέση με την απόδοση που έχουν. Ε, μπορεί πολλά να παίρνουν οι διαμεσολαβητές και λίγα οι, οι αποταμιευτές. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Επίσης, για να αποφύγω παρεξηγήσεις, θα πρέπει να πω ότι στην έκθεση υπάρχουν δύο κενά, πιστεύω εγώ. Καταρχήν, η χρηματοπιστωτική κρίση δεν ε, τέλειωσε ε, απλώς ε, διαφοροποιήθηκε. Αν δούμε τα επιτόκια βλέπουμε ότι έχουμε πολλές, ε, ε, πολλά κεφάλαια στις αγορές που δεν ξέρουν πού να επενδυθούν. Συμφωνώ με τον Φάμπιο Ντιμάζη που λέει ότι αυτό δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε με, με, με, με κάποιες επιπόλαιες ρυθμίσεις. Θέλουμε τα πλεονάσματα αυτά μακροπρόθεσμα να διοχετευθούν σε επενδύσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει στην έκθεση να κληθείτε ε, να δείτε ε, μακροπρόθεσμα το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προσέξετε ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν νέοι κίνδυνοι επειδή δεν θα γίνουν μακροπρόθεσμες αηφόρας επενδύσεις ε, που μπορεί να δημιουργήσουν νέους κινδύνους. Η διάσκεψη για το κλίμα ε, βεβαίως θα πρέπει να σας έδωσε τροφή για συμπεράσματα και σκέψη και τα περιμένουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κέινς είπε ότι αν χρωστάς σε μια τράπεζα 100 δολάρια έχει πρόβλημα, αν όμω χρωστάς ένα εκατομμύριο έχει αυτή πρόβλημα. Ή στην ε, κρίση ε, ε, οι τράπεζες, ε, ε, στις τράπεζες χρωστούσαν εκατομμύρια αλλά τελικά το πρόβλημα το είχαν οι πολίτες και η νομοθεσία μας έχει σκοπό να αποφύγει την επανάληψη αυτού του φαινομένου και ταυτόχρονα να αποφύγει την υπερβολική γραφειοκρατία που αυξάνει το κόστος των υπηρεσιών προσφέρων. Η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειώσει την νομοθεσία της είναι εξίσου αστεία με, το, με το, αυτό που λέγεται ότι η Βρετανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο και μόνο για το εμπορικό κομμάτι. Τελικά ε, πηγαίνουμε σε μια περισσότερη Ευρώπη με περισσότερο κόστος και περισσότερη γραφειοκρατία. Οι χρηματοπιστωτικές ε, εταιρείε ε, αντιλαμβάνονται ότι για να ξεφύγουν από το, τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μετακατασταθούν. Κύριε Μόνο. Κύριε Πίτροπε. Λυπάμαι που η έκθεση αυτή αγνοεί πολλά θέματα. Πρώτον, την ε, πραγματική τραπεζική ε, διαφοροποίηση και διαίρεση. Όλη η νομοθεσία ε, θα αποτύχει αν δεν διαχωρίσουμε τις τραπεζικές δραστηριότητες που έχουν μεγάλο κίνδυνο από τις υπόλοιπες. Γιατί αλλιώς θα παίζουν ρουλέτα τα χρήματα άλλων. Ε, οι πατριώτες αυτό ακριβώ καταγγέλουν ε, να, κάνει, να βγάλει κανείς ε, κέρδη με τα λεφτά άλλων όμως οι άλλες πολιτικές ομάδες και ιδιαίτερα το ΕΛΚ επιθυμεί τη διατήρηση της κατάστασης όπως έχει από την 1η του 2016 μάλιστα γίνεται ακριβώς το αντίθετο πηγαίνουμε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και βλέπουμε και το τα αποτελέσματα με τα τραπεζικά σκάνδαλα της ε, Ιταλίας. Δεύτερο θέμα, η τιτλοποίηση. Θα πρέπει να ανησυχούμε για ένα μηχανισμό που δημιούργησε κοινωνικά και οικονομικά, κοινωνικές οικονομικές μιας τεράστιας Πολιτεία. Είναι το κουτί της Πανδώρας. Τέλος, για την ε, Ένωση ε, Κεφαλαιογορών η... Δεδομένου ότι τα αιτήματα είναι μικρά, πολύ μικρά, η, ζήτηση είναι πολύ μικρή, οι επενδύσεις ε, δεν πρόκειται να επηρεαστούν από αυτή την ένωση θετικά ε, με κάποιο σημαντικό τρόπο. Ε, τελικά αυτό που θα γίνει είναι μετακίνηση στις Αμερικανικές τράπεζες και στα Αμερικανικά ιδρύματα που έχουν έδρα στο City. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στον Επίτροπο με μία ερώτηση. Ο νέος κανονισμός, αν δοθεί μέσα από το πρίσμα του καταναλωτή, ε, περιλαμβάνει τρία σημαντικά θέματα. Ενημέρωση, πολύ διεξοδική προς τον καταναλωτή, ε, ευθύνη τραπεζιτών, αναφέρατε και αυτό, ευθύνη και εποπτεία τραπεζών. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η τραπεζική εποπτεία να είναι στιβαρή και αποφασιστική. Και πάνω σε αυτή τη βάση σας ρωτώ, ξέρετε ότι στη χώρα μου, την Ουγγαρία, έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, και όχι μόνο στην Ουγγαρία μάλιστα, αλλά και σε πολλές άλλες ε, χώρες μέλη, ε, ε, λόγω των δανείων σε ξένο νόμισμα. Πολλοί άνθρωποι ε, προσελκύστηκαν και μπήκαν σε μια παγίδα για να πάρουν ένα δάνειο σε ξένο νόμισμα. Τώρα τι προσδοκίες έχουμε, γιατί μιλάμε τώρα για την ενημέρωση της σωστή των καταναλωτών και των υποψηφίων δανειοληπτών. Ε, θα πρέπει να... Γιατί, γιατί είναι αυτό κάτι καινούριο και καινοφανές, γιατί πιστεύετε ότι η Ευρωπα... τι, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ανθρώπους που είναι εκατοντάδες και που έκαναν λάθος και ε, έπεσαν στην παγίδα ε, και πήραν ε, δάνειο σε ξενονόμισμα. Ο κ. καλησπέρα σας. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Μπάλτση για αυτό το έγγραφο και να ε, ευχαριστήσω και τον κύριο Χίλ για την παρουσία του. Θα ελπίζω θα μας ε, βοηθήσει να προσανατολίσουμε τις ε, χρηματοοικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι έχουμε δύο σημαντικά project. Την Τραπεζική Ένωση που θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να κλείσει με την εγγύηση καταθέσεων και την Ένωση Κεφαλαίου που θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ε, αγορά κεφαλαίων, κεφαλαία αγορά της Ευρωζώνης ε, και να κινητοποιηθούν κεφάλαια σε νέα επενδυτικά σχέδια. Ε, δύο σημαντικές προτάσεις συζητώνται όμως και με ανησυχούν λίγο. Πρώτον, η ιδέα ότι χρειάζεται να ε, ε, αναθεωρήσουμε την ιδέα, να, ξανα, να επιστρέψουμε στην ιδέα ότι το, ε, το, το κρατικό χρέος θα είναι χωρίς κίνδυνο. δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή την ιδέα. Δεύτερον, η ιδέα ότι Έχουμε υπερβολική νομοθεσία για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Όχι, ε, θα πρέπει να δούμε βέβαια να βελτιώσουμε την νομοθεσία, ε, να δούμε που υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, αλλά όχι να λέμε ότι είναι υπερβολική η νομοθεσία και η ρύθμιση. Ευχαριστώ. Κύριος Λούνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό στο μέλλον το θέμα της αποταμίευσης. Όταν μια τράπεζα έχει προβλήματα, οι καταθέσεις προστατεύονται μόνο μέχρι 100.000 ευρώ. Στο μέλλον όμως θα πρέπει οι τράπεζες να επομιστούν αυτή την ευθύνη. Θα είναι οι, να είναι οι τράπεζες οι οποίες θα έχουν ένα μηχανισμό προστασίας. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε κατά πόσο στο μέλλον οι τράπεζες θα μπορέσουν να είναι ευφιέστερες με τη χρήση των καταθέσεων αυτών, <clears throat> των χρημάτων των καταθετών. Θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο στην Ευρώπη, όλες οι τράπεζες να συνεργαστούν για το εγχείρημα αυτό και να διευκρινίσουμε καλύτερα τι θα πρέπει να συμβεί. Θα πρέπει και οι τράπεζες του Βορρά να είναι αλληλέγγυες με τις τράπεζες του Νότου, τις τράπεζες της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη. Και εδώ είναι το θέμα πώς θα αποφύγουμε να υπάρξει μια τέτοια κατάσταση η οποία θα οδηγήσει σε διάχυση ευθυνών. Εγώ υπήρξα συγγητής για το θέμα αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ο κύριο Βέγγερς. Η κρίση του 2007 για ορισμένου, οφείλεται σε μια αποτυχία της ρύθμισης. Αυτό είναι λαθασμένη διάγνωση. Εμείς δημιουργούμε μια ψευδέστηση, να θεωρήσουμε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να αντιθασευστεί. <clears throat> ότι μπορούν τα συμφέροντα των τραπεζών και των hedge funds να ευθυγραμμιστούν με τα συμφέροντα των πολιτών και των εργαζομένων. Ένας μηχανισμός όπως ο μηχανισμός επίλυσης δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα όπως φάνηκε στην Πορτογαλία πρόσφατα όπου κρύφθηκαν πληροφορίες και διαστρεβλώθηκαν για να μην μπορούν οι ρυθμιστέ να ξέρουν περί τίνος γίνεται. Το πρόβλημα των τραπεζών που είναι too big to fail δεν μπορεί να λυθεί με μονάχα καταπραγητικές λύσεις, οι οποίες δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα μονάχα μπορεί να λυθεί με ένα δημόσιο έλεγχο του πιστοτικού ε, συστήματος για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την κρίση που αδύρυτα θα έρθει. Ευχαριστώ, ο Δεν βλέπω τον κύριο Μποργέτσιο. Ούτω, ως εκ τούτου δίνω το λόγο στην κυρία Γκέου. Mm. Mm. Καταρχήν συγχαρητήρια αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη ανάμεσα στην ε, βελτίωση της ε, πρόσφασης στη χρηματοδότηση και στην αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας και των ρυθμιστικών κειμένων μας. Ε, ε, μπορούμε, πρέπει να καλύψουμε τα κενά, αλλά όχι να υποχωρήσουμε ε, στις ε, ρυθμιστικές μας προσπάθειες. Θα πρέπει να μάθουμε από το αυτό που στην Κίνα. Πρέπει να διαθέτουμε ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να δια, διατηρήσουμε την ιδέα στο μυαλό μας. Η, επίσης, η Ένωση Κεφαλαιογορών δεν θα είναι πανάκια δεν θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, δεν πρόκειται να, ε, από μόνη της να βελτιώσει την ανάπτυξη, αλλά μπορεί να δώσει εναλλακτικέ ε, πηγές χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις ε, που σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, μόνο, και όχι μόνο σε επιχειρήσεις των χωρών που έχουν επιτυχημένες κεφαλαίες αγορές. Το ερώτημα είναι Μπορούμε να μιλούμε για ένωση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ε, ένα χώρο στον οποίο το κεφάλαιο να μπορεί να κινείται ελεύθερα χωρίς να παρεμποδίζεται από την εθνική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή όχι. Ε, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, Επίτροπε, γιατί αλλιώ ε, τα επενδυτικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελούν σταγόνα εν το ωκεανό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εθνικό κατακαιρματισμό επιγόντω. Ταυτόχρονα θα πρέπει οι μεσαίου, μεσαίους εταιρείε ε, να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση και αυτή η, ε, η, η, η, ρύθμισή μας, το ρυθμιστικό μας πλαίσιο θα πρέπει αυτό να το διευκολύνει, να επιτρέπει τι επενδύσει αυτές τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στο Catch the Eye, θα ήθελα να ζητήσω την συνεργασία σα έτσι ώστε να ε, τηρήσουμε τους χρόνους μας, το χρονικό μα ε, πλαίσιο, γιατί έχουμε καθυστέρηση. Επτά έχουν ζητήσει το λόγο, όμως ε, θα τον δώσω σε πέντε. κυρία Μάλετης, καταρχήν, λοιπόν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Χιλ στην Ολομέλεια και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μπάλτ, τον εισηγητή για την έκθεσή του. Χαιρετίζω τα μέτρα τα οποία προτείνονται σε αυτή την έκθεση. Τα αποδέχομαι και ιδίω την έννοια της ανάπτυξης της αγοράς γιατί αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κεφάλαιο. Πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμβάλλουν στο να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Επομένως, οι επιχειρηματίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε χώρες ιδίω όπου δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες κεφαλαίες θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις πιστοτικές αγορές στην Ευρώπη. Φυσικά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα και να εφαρμόσουν τις απαραίτητε διαρθρωτικέ αλλαγέ, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα του επιχειρήσεων στην Ευρώπη και οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω καλύτερων τρόπων χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Eh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συγγνώμη, αλλά δεν σας άκουσα να λέτε το όνομά μου. Με συγχωρείτε. Ε, συμφωνώ με την έκθεση που μας υποβάλλεται. Μετά από διεξοδική μελέτη καταλήγω ότι αντικατοπτρίζει σωστά την κατάσταση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Φαίνεται πόσο διαφέρει η κατάσταση μεταξύ Ευρώπης και ΕΠΑ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις, να φροντίσουμε ότι υπάρχει καινοτομία για τη βιομηχανία μας, για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Βέβαια, είναι αναγκαίο η πολιτική αυτή να μην, είναι, να μην δοθεί μόνο εργαλειακά, θα πρέπει να οδηγεί και σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και εδώ μιλάμε για τη ρυθμίση των αγορών. Δεν ε, συμφωνώ με κάτι που είπε ένας συνάδελφος από την αριστερά. Δεν υποστήριξε τη ρύθμιση των αγορών. Ε, παράλληλα όμως λυπάται διότι δεν είναι συγκεντρωτικό το τραπεζικό σύστημα. Αυτά τα δύο όμως ε, συμβαδίζουν. Τραπεζικών και άλλων συναλλαγών έχουν κομβικό ρόλο για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πολλάκις με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού και τα capital controls είναι ακόμη σε ισχύ οι αυξημένες χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες στις διατραπεζικές συναλλαγές επιβαρύνουν υπέρμετρα τους έλληνες χρεώσεις από 2 έως και πάνω από 10 ευρώ για απλή ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων για ποσά μέχρι 1000 ευρώ προμήθειες από 1 έως 1,25 ευρώ για πιστωτικές κάρτες προμήθεια στην τράπεζα της τάξης του 2 με 2,5% για μικρά και μεσαία εμπορικά καταστήματα ενώ αντίθετα για τα πολύ μεγάλα καταστήματα η προμήθεια είναι χαμηλότερη του 1% και όλα αυτά παρότι ο κανονισμός 751 ένα του 15 προβλέπει μεταξύ άλλων μέγιστες χρεώσεις για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μηδέν τριάντα και μηδέν είκοσι ευρώ αντίστοιχα. ταυτόχρονα οι τράπεζες καθυστερούν υπερβολικά την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων και εγγράφων τα οποία είχαν και έχουν ακόμη ανάγκη οι δανειολήπτες για κόκκινα δάνεια για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου κατσέλη για να γλιτώσουν τα σπίτια τους από τα κοράκια. αυτές οι πρακτικές των τραπεζών πρέπει να σταματήσουν και εσείς κύριε επίτροπε οφείλετε να λάβετε άμεσα μέτρα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε μια αγορά κεφαλε κεφαλαίου μια ένωση αγορών. Οι μας είναι σαφής. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στα δάνεια για τους καταναλωτές, έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι ορθά τεθειμένοι. Πρέπει όμως να βρούμε τον τρόπο να αντλήσουμε τα διδάγματα από τα σφάλματά μας, από τη χρηματοπιστωτική κρίση και ιδίως θα πρέπει να διδαχτούμε από αυτά τα οποία κάνανε στο παρελθόν οι τράπεζες προς τους πολίτες. Υπήρχαν αυτές οι απάτες που κάνανε οι τράπεζες. Σκεφτείτε όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι πήραν <coughs> δάνεια σε ελβετικά φράγκα. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα απατών. Ας τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας για το μέλλον. Ο κ. Σότς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η χρηματοπιστωτική κρίση ακόμα ε, είναι μεγάλη στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις της ορατές. Υπάρχουν θετικές και αρνητικές εξελίξεις ανάλογα με το που κοιτάμε. Πάντως οι πολίτες μας ε, δεν ε, είδαν μεγάλη βελτίωση και το ίδιο ε, ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα, την αλλαγή της νομοθεσίας όταν πρόκειται για χρηματοοικονομικές αγορές, όλα αυτά πρέπει να γίνουν πάνω στη βάση πολύ προσεκτικής ανάλυσης. Αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε μπροστά. Το ερώτημα είναι γιατί κάνουμε όλα αυτά τα βήματα. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε τον καταναλωτή, τον πολίτη, όχι μόνο τις τράπεζες και τους μεγάλους ε, οικονομικούς πρωταγωνιστές. Ε, ποιος θα εξυπηρετήσει με τις τράπεζες ή το, την πραγματικότητα των πολιτών μας. Ε, οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν πήραν το λόγο σύμφωνα με το άρθρο 162.12 ε, μπορούν να υποβάλουν ε, την παρέμβασή τους γραπτός υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνάει τις 200 λέξεις. Ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ε, ποικίλε παρεμβάσεις. Ε, αν εστιαστούμε καταρχήν στην έκθεση, πολλά από τα σχόλια ε, αναφέρθηκαν στην μοναδική θέση του χρηματοοικονομικού τομέα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, δεν είναι αυτός ο σκοπός, ε, είναι ένα μέσον για να πετύχουμε το σκοπό μας. Ε, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία της Ευρωπαϊκή Ένωση και προ όφελο όλη τη κοινωνία με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσει εργασία και να δοθεί στου πολίτε η σιγουριά να προγραμματίσουν το μέλλον τους ε, για όταν γεράσουν. Γι' αυτό το λόγο, κατόπιν της υιοθέτησης ε, ε, μια σειράς νομοθετημάτων ως αντιμετώπιση της ε, κρίσης, ε, ήταν σημαντικό και είναι σημαντικό, όπως λέει η έκθεση, να δούμε αν το σύστημα λειτουργεί όπως το είχαμε προβλέψει. Δεν θα ε, αμφισβητηθεί η βασική αρχιτεκτονική των μεταρρυθμίσεων, αλλά θα αναρωτηθούμε αν διατηρώντας την χρηματοοικονομική σταθερότητα ε, δεν παρεμποδίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει τέσσερα εργασίας και να παραμείνει ανταγωνιστική. Γιατί πολύ συχνά ε, σε τέτοιου είδους ε, ρυθμιστικούς ε, κανόνες, έτσι και εδώ, όπως ε, συχνά σε τέτοιους ρυθμιστικούς κανόνες, θα πρέπει να δούμε αν τηρούμε την ισορροπία. Το πρώτο βήμα ήταν η συλλογή πληροφοριών και αυτό θα λήξει σε 15 περίπου μέρες. η προσέγγιση δική μας είναι χωρίς προκαταλήψεις ε, οι πληροφορίες που θα πάρουμε θα μας επιτρέψουν να δούμε πώς λειτουργεί η νομοθεσία, ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα νομοθετικά και εθνιστικά κείμενα, αν υπάρχουν κενά, αν υπάρχουν επικαλύψεις Και πιστεύω ότι αυτές οι πληροφορίες θα είναι αρκετά λεπτομερείς έτσι ώστε να χτίσουμε την, οικοδομήσουμε την ανάλυση μας και τις συστάσεις μας. Όταν διαθέτουμε αυτές τις συστάσεις θα τις συζητήσω μαζί σας και θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εθνικά εμπόδια στα οποία αναφερθήκατε πολύ συχνά σήμερα και να οικοδομήσουμε μια πραγματική ενιαία κεφαλαγορά στην Ευρώπη. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, την ε, συνεισφορά τους που ήταν πολύ χρήσιμη. Έκλεισε το μικρόφωνο πάλι. Όλα αυτά είναι σημαντικά για όλους μας. Μετά από πέντε χρόνια νομοθετική εντατική δουλειά, μετά την αναδιάρθρωση σε οικονομικής εποπτείας και με προοπτική την Κεφαλαϊκή Ένωση και Ένωση Κεφαλαιαγορών, ε, ήρθε η ώρα να δούμε τον αντίκτυπο μέχρι τώρα και να ελέγξουμε μήπως ε, επιδέχονται όλα αυτά βελτιώσεις. Τα πρώτα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστά και οι τρέχουσες διαβουλεύσεις είναι με το, το, χρηματοπιστωτικό τομέα είναι θετικές. Οι διαβουλεύσεις ε, θα πρέπει όμως να λάβουν υπόψη και τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Επίσης η αναθεώρηση της οδηγίας CDI 4 είναι, έχει μεγάλο δυναμικό για απλοποίησης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ε, ωφελώντας έτσι κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εννοώ εδώ. Ε, σίγουρα ε, μια πρόοδος εδώ είναι σημαντική. Ως Επιτροπή ΕΚΟΝ ζητούμε σωστά να, σε τακτά διαστήματα να γίνεται μια εξέταση της αναλογικότητας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Τονίζω επίσης κύριε Επίτροπε ότι στη μελέτη του αντίκτυπου ε, δεν πρόκειται μόνο για ε, ε, ένα μόνο κομμάτι αλλά για ένα γενικότερο πλαίσιο. Έτσι θα δούμε τις αλληλεξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις και με αυτόν τον τρόπο θα είναι λιγότερο σύνθετες οι διαδικασίες και οι στόχοι θα εφαρμοστούν καλύτερα. Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει την ε, υποχρέωση να αναλάβει πρωτοβουλία. Επίση, οι εποπτικές αρχές και η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να φροντίσουν για τη βελτίωση όλων αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να παραμείνουν πρακτικές και αναλογικές. Η ποιότητα και η τήρηση των νόμων θα πρέπει να αντιμετωπίζετε ξανά ως προτεραιότητα. Για το έργο σας σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κλείνει η συζήτηση, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης.